Uh, παρακαλώ στις θέσεις σα, παρακαλώ στη θέση σα και καλώ ήρθατε στη σημερινή απογευματινή συνάντησή μα. Um, Ζητώ συγγνώμη, η αίθουσα δεν είναι αρμόζουσα. Δεν μπορέσαμε να βρούμε μια άλλη αίθουσα για αυτούς που θέλουν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση. Ζητώ συγγνώμη, προσπαθήσαμε παρόλα αυτά. Αν μπορείτε όμως, καθίστε, όσοι πρέπει να βγείτε, βγείτε, για να αρχίσουμε. Η κυρία Ρούλε, η οποία είναι η εισηγήτρια για τον προπολογισμό βάσει της νέας διαδικασίας, θα ήθελε να πάρει το λόγο σύντομα, γιατί ακριβώ δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, για να μας μιλήσει για κάποια θέματα τα οποία πρέπει να αναφερθούν σήμερα. Πρόκειται για μια νέα διαδικασία. Κυρία Ρούλε, έχετε το λόγο. Ναι, ναι, θα είμαι πάρα πάρα πάρα πολύ σύντομη. Όπως ξέρετε, βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας, σας παρακαλώ σιωπή, λέει ο Πρόεδρος. Αποκτήσαμε σαν κοινοβούλιο, συνεχίζει η κυρία Ρούλε, νέες αρμοδιότητες και νέα δικαιώματα. Υπάρχει σήμερα η πρώτη ανάγνωση, η μία και μοναδική ανάγνωση και επαναλαμβάνω το κοινοβούλιο έχει νέα δικαιώματα, νέες αρμοδιότητες. Ακριβώς επειδή η Επιτροπή καθυστέρησε δεν έχει πλέον τη δυνατότητα για το 2011 να υποβάλει τις κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό λοιπόν θα το κάνει το Κοινοβούλιο. Είμαστε οι πρώτοι που θα γνωμοδοτήσουμε, οι πρώτοι που θα πάρουμε θέση και πρέπει να το κάνουμε σχετικά γρήγορα. Στι 4 Μαρτίου, όπω ξέρετε, θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμού. Εμεί λοιπόν εδώ, σαν δική μα Επιτροπή, σαν Επιτροπή Εσωτερική Αγορά, αν θέλουμε να υποβάλουμε κάποιε προτάσει, πρέπει να το κάνουμε μέσω των συντονιστών. Σήμερα θα υποβάλω την επιστολή στους συντονιστές με τις δικές μας κατευθυντήριες γραμμές, τις δικές μας οδηγίες και θα ζητήσω από τους συντονιστές για να τηρηθούν οι προθεσμίες να ακολουθήσουν την διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα. Αλλιώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε θέση. Πρόεδρος, σήμερα το απόγευμα αργότερα θα συνεδριάσουν οι συντονιστές. Έχετε δίκιο να ενημερώνετε όμως και όλα τα μέλη της Επιτροπής. Οι συντονιστές θα επιληφθούν του σήμερα το βράδυ. Πρόεδρο, σας παρακαλώ, αν δεν έχετε θέση, δεν μπορώ να δεχτώ όρθιους εδώ, οι οποίοι κουτσομπολεύουν. Ζητώ συγγνώμη, αλλά θα πρέπει ε, να βγείτε από την αίθουσα Ζητώ συγγνώμη αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για όλους, αρκετές θέσεις. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αν δεν υπάρχει ησυχία μέσα στην αίθουσα. Και δυστυχώς δεν έχουμε ε, αίθουσα για αυτούς που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν. Σας παρακαλώ πολύ όμως όλοι όσοι είστε όρθιοι να παραμείνετε σιωπηλοί. Προχωρούμε στην πρώτη ψηφοφορία. Θα χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες, όχι συνέχεια, απλώς εάν η ε, ψηφοφορία το απαιτεί, αν το αποτέλεσμα είναι αμφίβολο. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν, θα ήθελα στην αρχή να ελέγξουμε το σύστημα Εντάξει. Ποιος ψηφίζει για το ΕΛΚ παρακαλώ. Ελέγχουμε. Όχι κυρία Γκέφχαρτ, ναι το ξέρω. Ποιος ψηφίζει για το ΕΛΚ παρακαλώ πολύ ψηφίστε τώρα για να δούμε και να μετρήσουμε. 14 ψήφους έχετε μόνο. Κάτι λάθος έγινε. Κάποιος πρέπει να βγάλει την κάρτα του για να φτάσουμε στον αριθμό 14. ΕΛΚ. Είμαστε στο 16. Δύο πρέπει να βγούνε. 17. Από το 16 πήγαμε στο 17. Όλο και περισσότεροι ψηφίζουν για το ΕΛΚ. Κάτι δεν πάει καλά. 16. Δεν μπορούμε να περιμένουμε όλη τη μέρα. Σας παρακαλώ πολύ. Δύο άτομα δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. 14 μόνο. Όχι, τώρα πήγαμε στο 13. 13 ή δεκατέσσερις, αλλά όχι παραπάνω. Εντάξει. Το ΕΛΚ λοιπόν 14. SND. Κυρία Γκέπχαρτ. Οι σοσιαλιστές. 10. Ωραία. Τέλεια. Άλντε. Άλντε παρακαλώ πολύ. Έλεγχος. Δύο. Μόνο δύο. Όχι. Τέσσερις. Ωραία. Η πράσινη. Δύο. Τρεις. SDR. Εγώ δεν ψηφίζω. Δύο ή τρεις. Γκουέ. Κύριε Τριανταφύλλου. Δύο. Δύο. Ναι, μπορείτε να ψηφίσετε κυρία Στάσεν. Ποιος άλλος. Δύο. Μία εγγεγραμμένη. Εντάξει. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, η συγχύτρια. Γρήγορα, γρήγορα, πολύ γρήγορα. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την πολύ καλή συνεργασία μαζί τους. Εντάξει και για το τελικό αποτέλεσμα να δούμε τι θα γίνει, αλλά ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες οι οποίοι βοήθησαν, προσπάθησαν, ασχολήθηκαν με αυτό και κάτι το θετικό ότι πάρα πολλοί προσπάθησαν ε, για να δουν ε, τι θα γίνει με τις ετικέτες των τροφίνων μας στο μέλλον. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και ευχαριστώ και πάλι. Εντάξει, υπήρξαν ε, και κάποιες συμβαστικές τροπολογίες, κάτι που διευκολύνει την Ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 119, 110 καταπίπτουν. Περνάμε στην επόμενη υπέρ. Α, εδώ χρειάζεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. 19 υπέρ, 17 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στο 2. Όλες οι τροπολογίες από πέντε διαφορετικές πολιτικές ομάδες, πιστεύω ότι θα ψηφίσουμε από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 μάλλον 11 11 11-12 καταπίπτουν και περνάμε στην παράγραφο 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα περάμε στην προφορική τροπολογία 2. Υπέρ, ναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται έλεγχος. Και περνάμε στην 13 της κυρίας Σάλτε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 3. Παράγραφος 3, 115 του κυρίου Κάρας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δύο τροπολογίες, η 14 και η 114, Ντεγιόν και Σάλτεμόζα. Ποιος είναι υπέρ. Νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε για τη 14 και την 114. Τέλος. Απορρίπτεται. 21 υπέρ, 15 κατά μία εποχή. Και τώρα περνάμε στην 116 της κυρίας Μακάρτη υπέρ Ηλεκτρονική ψηφοφορία 116 της κυρίας Μακάρτη. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται 21 υπέρ 15 κατά χωρίς αποχές. Άρθρο 4. Εδώ έχω ένα πρόβλημα. Όταν ψηφίζω ναι, μου λέει όχι και όταν... Ε, μου κάνει τα αντίθετα τέλος πάντων το μηχάνημά μου. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που είναι υπέρα η ομάδα σας και πέρασε η ψηφοφορία δεν υπάρχει θέμα. Περνάμε τώρα στο άρθρο 4. Δεν πειράζει κύριε. Περνάμε στην 117. Πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 117 ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται η 117, 29 κατά, 8 υπέρ, χωρίς αποχές. 118 της κυρίας Μακάρτη. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Υπάρχουν αποχές. Απορρίπτεται. 7 Άρθρο 7. Συμβαστικές τροπολογίες. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119, 120. 121 καταπίπτουν. 122 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 8. Τροπολογία 15 της κυρίας Αλταμόζα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. 123, Μακάρτη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 124 της κυρίας Ντεγιόγκ, υπέρ, Κατά. Εγκρίνεται. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 Σαλτεμόζα. Υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 16. Αρχή της ψηφοφορίας για τη 16. Τέλος. Εγκρίνεται. 17. Σάλτε Μόζα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. 17 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, 20 και κατά, χωρίς αποχές. 125 καταπίπτει, γιατί είναι προσθήκη. 18. Ψηφίζουμε την τροπολογία 18. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 18. Τέλος. 18. Υπέρ 18 κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε στο άρθρο 9 και την τροπολογία 19 της κυρίας Αλδεμόζα. Υπέρ ηλεκτρονική ψηφοφορία. 19. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Τέλος. Εγκρίνεται. 23 υπέρ 14 κατά. 126 κάρας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Σάλτε Μόζα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 δεν ψηφίζουμε είναι γλωσσική δύο παρόμοιες η 21 και η 128 Σαλντεμόζο και Κάρας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 της Σιγήτριας. υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συμβιβαστικές τροπολογίες. Τρία. Πέντε πολιτικές ομάδες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 131, 134, 130, 132 και 133 καταπίπτουν. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και μετά περνάμε στην 134, σβήνουμε ένα τμήμα μιας φράσης του κ. Αγγελιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στο άρθρο 10 και την τροπολογία 23 ηλεκτρονική ψηφοφορία. 10. Συγγνώμη, τροπολογία 23, άρθρο 10. Τέλος. 23 υπέρ, 14 κατά. Εγκρίνεται. 135. Η κυρία Μακάρτη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 24. Τροπολογία 24 της εισηγήτριας. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. 24. Αρχή της ψηφοφορίας. Αρχή. Τέλος. 21 υπέρ, 14 κατά, 2 εποχές. Άρθρο 13, 136 τροπολογία, De Young ηλεκτρονική ψηφοφορία. 136. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. 25 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. 14. Γίνεται ξεχωριστή ψηφοφορία. 139, De Jong. Βλέπετε στον κατάλογο που έχετε μπροστά σας πώς ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος του 139. Υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα του 139. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στην προφορική 3. Εάν δεν περάσει αυτό, όλα τα υπόλοιπα για το άρθρο 14 καταπίπτουν. Προφορική τροπολογία 3 λοιπόν. Συμφωνείτε? Συγγήτρια, ναι. Προφορική τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Προφορική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27-33 καταπίπτουν. 28. Τροπολογία 28 της εισηγήτριας. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της 28. Αρχή. Τέλος. Εγκρίνεται. 20 υπέρ, 18 κατά, χωρίς αποχές. 144. Έγκελ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 145. Λιόν. 145. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 146 De 146 Υπέρ Κατά Αποχές Απορρίπτεται 29 της εισηγήτριας Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 29 Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. 15 υπέρ, 23 κατά. 147 σαράντα επτά καταπίπτει. 147 καταπίπτει. Ψηφίζουμε λοιπόν την 147. 147 ψηφίζουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15, άρθρο 15. 149. υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 149. Τέλος. 19 υπέρ, 19 κατά. Απορρίπτεται. Κρίμα, κύριε Δε 150, τροπολογία 150, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 151 στο άρθρο 16, Σμιτ, υπέρ, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την 151. Τέλος. Εγκρίνεται. 19 υπέρ, 2 κατά, 2 εποχές. Άρθρο 17, 152, τροπολογία της κυρία Τεγιόγκ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Κύριος Διόγκ. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται 15 υπέρ 23 κατά. Χωρίς αποχές. Και περνάμε στην 153. Κάρας υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Δεν βλέπω κανέναν να θέλει να απέχει, γι' αυτό και δεν ζητώ αποχές, αλλά αν θέλετε πρέπει να το πείτε. Περνάμε στην παράγραφο 2, 154, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η επόμενη τροπολογία του κυρίου Κάρας καθώς και 156 καταπίπτουν και περνάμε στην 157 υπέρ κατά απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην 158 ε, Μακάρτιν υπέρ κατά εγκρίνεται. 30. Τροπολογία 30 καταπίπτει. Τώρα πάμε στη συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 159, 160 καταπίπτουν και πάμε στο άρθρο 20, 22. Τροπολογία 20, 32, συγγνώμη. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 32. Τέλος. Απορρίπτεται. 12 υπέρ 26 κατά. Και τώρα περνάμε στην 164, 165. Είναι Έγκελ και Μακάρτιν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 163, De Jong, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η επόμενη τροπολογία αποσύρθηκε. Και τώρα ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο, το άρθρο 20, με χωριστή ψηφοφορία, όπως ζήτησε το ΕΛΚ. Βλέπετε το αρχικό κείμενο, το πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα. Μάλλον θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι κα... υπέρ. Κατά. Βλέπω ότι υπάρχει ομόφωνη αντίθεση. Δεν υπάρχουν αποχές, οπότε είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άρθρο 21. 167 του κυρίου Κάρας. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 168 Κάρας. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται και αυτό. 22, άρθρο 22, 33, τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συμβιβαστικές τροπολογίες 5, Μπίλτ και Ριό. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 170 καταπίπτει. Ε, τώρα περνάμε στο άρθρο 24. 34 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25, άρθρο 25, 171, De Jong, υπέρ, ηλεκτρονική ψηφοφορία. 171 ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται 21 υπέρ 17 κατά, χωρίς αποχές. Και περνάμε στο άρθρο 29. 173 κάρας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 172 της εισηγήτριας Νομίζω πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 172. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. 172. 19 υπέρ 17 κατά δύο εποχές. 35 της εισηγήτριας. Υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. 35. Ψηφίζουμε την 35. Τέλος. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 5. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Εξού και περνάμε στην 37 της εισηγήτριας. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Νομίζω ότι η τροπολογία 17 καταπίπτει και περνάμε στην 38 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τη τροπολογία 38. Τέλος. Απορρίπτεται. 17 υπέρ 21 ψήφους κατά. 178, τροπολογία de υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία Engel που θα ψηφίσουμε σε δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες. Πρώτο τμήμα, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας του κριμά Engel. Υπέρ. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 23 υπέρ, 14 κατά. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η επόμενη τροπολογία Build 180 καταπίπτει το αρχικό κείμενο επίσης και περνάμε στην τροπολογία 182 κάρας υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 183 Μακάρκιν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η επόμενη τροπολογία είναι η τροπολογία Μπατ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 40 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές Α, η 41 καταπίπτει. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. 184 είναι η επόμενη. 184, παράγραφος 3, Μακάρκιν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Παράγραφος τροπολογία 42 της συγκήτρης, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Άρθρο 30. Έχουμε την τροπολογία Κάρας 185 με δύο διαφορετικές ψηφοφορίες. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικό της έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας του κ. Κάρας. Κάντε πιο γρήγορα παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται 21 υπέρ 17 κατά. 31, άρθρο 31, συμβιβαστική τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά αποχές εγκρίνεται. Πολλές τροπολογίες καταπίπτονται, θα τις διαβάσω όλες, αλλά πάμε στην 196 Κρόιτσμαν 2α Άρθρο 31 Ποιος είναι υπέρ 196 κατά αποχές απορρίπτεται Προφορική τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Προφορική 6. Υπέρ. Αρχικά το είχε υποβάλει το ΕΛΚ και τώρα είναι κατά. Κατάλαβα καλά, λέει ο πρόεδρος. Προφορική τροπολογία 6. Τώρα το ΕΛΚ είναι κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ναι, δικαίωμά σας. Η ομάδα του ΕΛΚ θέλει πραγματικά να απορριφθεί η δική τους τροπολογία. Ψήφισαν 39. Απορρίπτεται. 16 υπέρ, 19 κατά. Δύο ποχές. Αυτό σημαίνει ότι ψηφίζουμε την τροπολογία 44 της εισηγήτριας. Γιατί δυστυχώς δεν πέρασε η προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία της εισηγήτριας. Τέλος. Απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά. Περνάμε στην τροπολογία Τέρμεν. Ηλεκτρονικά. 198 είναι η τροπολογία αυτή. Πολύ αργά ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 10 υπέρ 24 κατά. 201. Τροπολογία Λιό. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. «201» είναι η τροπολογία. Τέλος. Απορρίπτεται. 7 υπέρ, 30 κατά. Άρθρο 31. Παράγραφος 3. 202. Κρόιτσμαν και Βάισκεμπ. Ένα διαδικαστικό κύριε Πρόεδρε έχω. Έχουμε βγάλει τη λέξη mandatory υποχρεωτικά και έχουμε βάλει τη λέξη voluntary εθελοντικά και το ρήμα shall στη θέση του may. Αναφερόμαστε λοιπόν στα διάφορες προσθετικέ ουσίες, αλάτι, ζάχαρη κτλ. τα Κατά κάποιο τρόπο στη φράση αυτή είναι η λογική συνέπεια αυτού που λέμε. Είναι προφορική η τροπολογία σας, θέλετε να την υποβάλλετε. Μπορώ να το δεχτώ μόνο αν οι πολιτικέ ομάδες το δέχονται. Η εισηγήτρια καταρχήν. Συμφωνείτε. Υπάρχει κάποιος που έχει αντίρρηση σε αυτή την προφορική τροπολογία. Πρέπει να το ξανακούσουμε για να κατανοήσω περί τίνος πρόκειται. Εδώ προτείνουμε να πάμε από υποχρεωτική δήλωση σε εθελοντική δήλωση. Η λογική συνέπεια εδώ σε αυτή τη φράση είναι να αντικαταστήσουμε το shall με may. values, energy content, fat, saturated sugars and salt may in addition be expressed as appropriate a percentage of the reference intakes and so on. Is everybody happy with that? Okay. Right. So I put then amendment 202. Όπως τροποποιείται προφορικά, τώρα το θέτω σε ψηφοφορία. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. 202 όπως τροποποιήθηκε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 έναντι 8 με 10 αποχές. Οπότε η 199 καταπίπτει όπως και η 200. Προχωρούμε λοιπόν στη 203 της κυρίας Τούρουνεν. Θέτουμε σε ψηφοφορία τη 203 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 32. 204 των Βάις Γκέρμπερ και Κρόιτσμαν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Καταρρύπτ. Απορρίπτεται. 205 της κυρίας Τουρούνεν. Ποιοι είναι υπέρ. Νομίζω ηλεκτρονικά θα το ελέγξουμε. 205 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 13 υπέρ, 24 κατά, 2 αποχές. Τροπολογία 186, Χοάνγκ Γκόγκ, ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές, καταρρίπτεται. 187 του κυρίου Κάρας. Ποιοι είναι υπέρ. Μπορούμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Την 187. Αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 23 έναντι 15 ψήφων χωρίς αποχές. Στην οποία περίπτωση 188 και 45 καταπίπτουν. Και περνούμε τώρα στον παράγραφο 2 του άρθρου 32. Τροπολογία 206. για τη σχετική απάλληψη της κυρίας Τουρούνεν. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, καταρρύπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 46. Σωστά, της κυρίας Σάλντε Μόζε. Ποιοι είναι υπέρ, Ηλεκτρονικά. Τροπολογία 46. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 19 έναντι 19 ψήφων. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 208 της κυρίας Κόμη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Επομένως οι 207 και 209 απορρίπτονται και περνάμε στην τροπολογία 47. Η 47 της κυρίας Σάλντεμόζη υπέρ ηλεκτρονικός έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 21 ψήφι έναντι 17. Μετά η 210 του κυρίου Χόανγκ Γκόγκ. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 210. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχισε η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 12 υπέρ και 27 κατά. Άρθρο 33. Τροπολογία 211 του κυρίου Κάρας. Ποια είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 212 των Βάις Γκέρμπερ Κρόιτσμαν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 21 έναντι 18. Άρθρο 34. Συμβιβαστική τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Στην οποία περίπτωση περνούμε στην τροπολογία 216. Άρθρο 34 παράγραφος 1α. Τροπολογία 216 λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 218. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49 της κυρίας Μόζε. Μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. 19 έναντι 19 ψήφων, επομένως απορρίπτεται. Στη συνέχεια περνούμε στην τροπολογία 50, de ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 50. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 έναντι 18 χωρίς αποχές. Τροπολογία 219 της κυρίας Κόμη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 217 του κυρίου Κρόιτσμαν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δύο ταυτόσιμες τροπολογίες, η 51 Σαλ και η 220 του κυρίου Ντε Αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 15 υπέρ, 24 κατά. Τροπολογία 221 του κυρίου Κάρας. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 222 της κυρίας Μακλάρκιν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52 της κυρίας Σάλντε Μόζε. Ποιοι είναι υπέρ. Μπορούμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 52. Πέρας της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24 ψήφοι έναντι 15. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 53 της εισηγήτριας. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 53. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 24 κατά. 15 υπέρ. Τροπολογία 223 των Βάις Γκέρμπερ Κρόιτσμαν. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 224 Κάρας. Ποιοι είναι υπέρ? Α, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Η 224. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 23 κατά 15 υπέρ. Απορρίπτεται. Ε, η 225 τώρα του κυρίου Κρόιτσμαν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 35. 226 του κυρίου Κάρας υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 227 της κυρίας Μακλάρκιν υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 228 του κυρίου Κρότσμαν υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 229. Ας το δούμε ηλεκτρονικά των κυρίων Ζουβέν Αμπάντ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 20 υπέρ 19 κατά. Ε, νομίζω αυτό σημαίνει ότι η 54 απορρίπτεται. Περνάμε στην ε, Καταπίπτει μάλλον. Περνάμε στην τροπολογία 55 της εισηγήτριας. Ηλεκτρονικά θα το κάνουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 55. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 55. Μάλιστα, είσαστε υπέρ. Ηλεκτρονικά θα το ελέγξουμε ούτως ή άλλως. Ναι, η 54 κατέπεσε, η 55. Ποιοι είναι υπέρ? 34 υπέρ, 5 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 230. Νομίζω ηλεκτρονική. 230 τον κύριο Ζουβέν και Αμπάντ. Μπορούμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 230. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 20 έναντι 19 ψήφων. Τροπολογία 56 της κυρίας Σάλντε Μόζε. Νομίζω ηλεκτρονικά και αυτό. 56 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 έναντι 23. Η 200... Συγγνώμη, απορρίπτεται. 231 καταπίπτει και περνάμε τώρα στο άρθρο 6 Τροπολογία 232 του κυρίου Κάρας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Κύριος Κάρας, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 έναντι 17 ψήφων. Από ότι όλες οι τροπολογίες για το κεφάλαιο 6 καταπίπτουν, γιατί ολόκληρο το κεφάλαιο διαγράφεται. Επομένως, περνάμε στην 229, αν δεν κάνω λάθος, στο κεφάλαιο 7. Αυτό είναι αρκετές σελίδες ε, αργότερα. Όλες οι τροπολογίες αυτές καταπίπτουν, σωστά. Έτσι δεν είναι, κύριε Σόλτεμος. Είμαστε στο κεφάλαιο 7. 2.29 του κυρίου Κάρας, 51 ε, του κυρίου Άμπαντ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνονται 19 έναντι 18 ψήφων. Αυτό σημαίνει ότι διαγράφονται τα επόμενα κεφάλαια, το 8, Οπότε πού πάμε τώρα στη 251. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι επόμενες τροπολογίες, αφού κατέπεσε το κεφάλαιο 7, δεν έχουν νόημα. Επομένως, περνάμε στην τροπολογία 251 του κύριου Κάρας. Άρθρο 53 λοιπόν. Τροπολογία 251. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ναι. Τροπολογία 68 της εισηγήτριας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά για την 68. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 20 ψήφοι έναντι 16. Περνούμε στην 252. Σωστά. 252 της κυρίας Βάις Γκέρμπερ σε δύο κομμάτια, δύο τμήματα. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της, δια... της 252. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το πρώτο μέρος της τροπολογίας 252. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 10 υπέρ 26 κατά. Αυτό σημαίνει ότι το δεύτερο καταπίπτει νομίζω. Ψηφίζουμε και το δεύτερο μέρος. Ψηφίζουμε και το δεύτερο μέρος. Ναι, ψηφίζουμε και το δεύτερο μέρος λοιπόν. Ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 252 της κυρίας Βάις Γκέρμπερ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 23 έναντι 15 με μία αποχή. Περνάμε στην τροπολογία Λιών 253 που επίσης είναι σε τμήματα χωριστή ψηφοφορία. Θέτω σε ψηφοφορία το πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Το δεύτερο της 253. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Πέντε υπέρ, 33 κατά. απορρίπτεται. Περνούμε στην... Μάλλον η 69 καταπίπτει. Περνούμε στο παράρτημα 1. Τροπολογία 254 του κυρίου Κάρας. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 255 της κυρίας Βάισγκέρμπερ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Ε, πανηγυρικά απορρίπτεται. Δεύτερο παράρτημα της κυρίας Μακλάρκιν, από τροπολογία 256. Ποιοι είναι υπέρ, Κατά. Απορρίπτεται. Παράρτημα 3. 258 της, Κυρίου της εισηγήτριας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 259 του κυρίου Κάρας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 70 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 257 της κυρίας Μακλάρκιν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στο παράρτημα 6, είπε ο πρόεδρος. Ε, τροπολογία 264. Είναι το παράρτημα 4. 264 άρχεται η ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. 264 πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24 ψήφοι έναντι 15. Κύριε Κάρας, καλά τα πάτε με τις τροπολογίες σας. Τροπολογία 72 της εισηγήτριας. Ποιοι είναι υπέρ? Α, συγγνώμη. Οι 72, οι 267 και 73 καταπίπτουν. Περνάμε στην τροπολογία 260 του κυρίου Κρόιτσμαν. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 261 και 265 των Βάις Γκέρμπερ και Κάρας, ταυτόσιμες τροπολογίες. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Απο... Απορρίπτονται οι δύο αυτέ τροπολογίες. Τροπολογία 262 του κυρίου Ντε Ιόγκ. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά? Απορρίπτεται. Τροπολογία 268 των Τιούν και Χόχενστάιν. Υπέρ? Νομίζω ηλεκτρονικός έλεγχος. Η 268. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 ψήφι έναντι 18 η 74 καταπίπτει και περνούμε στη 263 της κυρίας Γκέρμπερ. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 266, 263. Καλά, εντάξει, ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για τη 263. Πέρας τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 έναντι 17 ψήφων. Η 266 του κυρίου Κάρας. Ποιος είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Απορρίπτεται. 269 της, των Τουν και Χόχενστάιν. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Απορρίπτεται. Συγγνώμη κυρία Τούν. Τροπολογία 75 της εισηγήτριας. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Εγκρίνεται. Παράρτημα 5. Τροπολογία 76 της Σάλτε Μόζε. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Εγκρίνεται. επόμενος καταπίπτει 270. Περνάμε στο παράρτημα 6. Ήρθαμε στο 6. Τροπολογία 77 της Σάλτε Μόζε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78 της Ιδίας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στο παράρτημα 8. Τροπολογία 271 του κυρίου Κάρας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 272 της κυρίας Μακλάρκιν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η κυρία Βάισγκαρπερ. Ακούστε, Σχετικά με τις απομιμήσεις ε, για το 270 εκεί υπήρξε και ένα λάθος στο παράρτημα 5 γιατί το 270 θα έπρεπε να το ψηφίσουμε. Ακούστε. αν δεν είχε θετηθεί η συμβαστική λύση δεν έπρεπε να ψηφιστεί, αλλά πρέπει να ψηφιστεί. 270. Ένα θέμα πάνω στο οποίο συμφώνησαν όλες οι ομάδες είναι η ετικέτα για αυτά τα προϊόντα. Ναι, με σύμφωνα με τον κατάλογο ψηφοφορίας και ο εισηγητής τον είχε αποδεχτεί αυτόν τον κατάλογο ψηφοφορίας. Εντάξει, θέλετε να ψηφίσουμε, εντάξει. Ωραία, θα επανέλθουμε. Θα ψηφίσουμε την τροπολογία 270 της κυρίας Βάισγκαρμπερ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Πού ήμασταν. 273 της κυρίας Μακ Κλάρκιν, δεύτερη τροπολογία της κυρίας Μακ Κλάρκιν. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 79 της κυρίας Σάλντε Μόζε. Ποιοι είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Η κυρία Κρόιτσφελτ απέσυρε τη δική της, οπότε περνούμε στο παράρτημα 11. Ελπίζω να έχω δίκιο. Τροπολογία 275 του κυρίου Κάρας. Αρχίζει ηλεκτρονικά η ψηφοφορία για την 275 του κυρίου Κάρας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 23 έναντι 16 ψήφων. Τροπολογία 276 του κυρίου Κάρας. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Περνούμε στο παράρτημα 12, τροπολογία 277 του κυρίου Κάρας. Ποιοι είναι υπέρ? Ηλεκτρονικά παρακαλώ, επί της 277. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 έναντι 14, 14 ψήφων με δύο αποχές. Περνούμε στο παράρτημα 13. Τροπολογία 278 του κυρίου Κάρας. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 279 της κυρίας Μακλάρκιν. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 280 της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ. Ποιοι είναι υπέρ, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τροπολογία 280, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14 υπέρ, 25 κατά. Τροπολογία 281 του κυρίου Κάρας. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 282 των Βάις Κέρπερ και Κρόιτσμαν. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ επί της 282. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 έναντι 17 ψήφων. Περνούμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Ε, αιτιολογική σκέψη 10, τροπολογία 1 της κυρίας Σάλτεμόζε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 80, De Jong. Χωριστή ψηφοφορία έχει ζητηθεί εδώ. Αρχίζει η ψηφοφορία λοιπόν ηλεκτρονικά για το πρώτο τμήμα της 80. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 20... 21 έναντι 17 ψήφων με μία αποχή. Τώρα το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 80 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 4 υπέρ, 37 κατά, μία αποχή. Τροπολογία 81, Κρόιτσμαν. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2, της εισηγήτριας. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 72, De Jong. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, Μόζε. Υπέρ. Α, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Τροπολογία 3 της κυρίας Σάλτεμόζε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τελείωσε η ψηφοφορία εγκρίνεται 24 έναντι 15 ψήφων. Περνούμε στη συμβιβαστική τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, εγκρίνεται. Επομένως, περνούμε όλες οι άλλες τροπολογίες για την αντιολογική σκέψη 25 καταπίπτουν. Η Περνούμε λοιπόν στην τροπολογία 87 της κυρίας Μακλάρκιν. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 88 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 της εισηγήτριας. Παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τροπολογία 5 της κυρίας Μόζε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12 υπέρ 26 κατά μία αποχή. Έχουμε τώρα την 89 της κυρίας Τούρενεν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12 υπέρ 26 κατά. Περνάμε τώρα στην προφορική τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 28. Τροπολογία της κυρίας Αλντεμόζε. Ποιοι είναι υπέρ. Ηλεκτρονικά θα το ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 6. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12 υπέρ 26 κατά. Αυτό σημαίνει ότι η 90, είμαστε στην 90 τώρα της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 28 έναντι 16 ψήφων. Καταπίπτει επομένως η τροπολογία του κυρίου Ντεγιόγκ. Τροπολογία 92 της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 92. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 34 ψήφοι υπέρ, 3 κατά. Τροπολογία 93 της κυρίας Μακλάκιν. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 94 του κυρίου Ντεγιόγκ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 7 της κυρίας Σάλντομόζ. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 7 της κυρίας Σάλντομόζ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12 υπέρ, 27 κατά. Τροπολογία 95, Χοχ, Ποιοι είναι υπέρ. Νομίζω ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 95. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 12 υπέρ, 27 κατά. Αιτιολογική σκέψη 36, τροπολογία 96, De Jong. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 96. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 26 εναντί 13 ψήφων. Περνούμε λοιπόν τώρα στη συμβιβαστική τροπολογία 9. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και επομένως όλες οι άλλες τροπολογίες για την αιτιολογική σκέψη 37 καταπίπτουν και περνάμε στην 103 της κυρίας Κοράτσα Πίλτ. Τροπολογία 103. Αρχίζει η ψηφοφορία. Για την 103. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 έναντι 18 ψήφων. Έχουμε ε, μια νέα αιτιολογική σκέψη της κυρίας Αλντεμόζε. Τροπολογία 9. Αρχίζει η ψηφοφορία. Για την τροπολογία 9. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 15 υπέρ, 22 κατά, 2 αποχές. Μετά, αιτιολογική σκέψη 39, τροπολογία 104 της Κοράτσα Μπίλτ. Αρχίζει η, πλειούς, η, ψ, η ψηφοφορία. Την αποσύρατε. Ωραία. Περνάμε στην συμβιβαστική τροπολογία 10. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Γι' αυτό περνάμε τώρα στην ε, τροπολογία 107 του κυρίου Κρόιτσμαν. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. Και τελική τροπολογία 108 του κυρίου Κρόιτσμαν. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται. Πριν περάσουμε στην τελική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης συνολικά, θα δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια για να πει λίγα λόγια. Κυρία Σάλντο Ναι, λυπάμαι που θα πρέπει τώρα να λάβω το λόγο αυτή τη στιγμή της ψηφοφορίας, αλλά να σας πω ότι μετά από το αποτέλεσμα του 6 και του 7, και του 7 θα έπρεπε να δούμε αυτή τη δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν και συμπληρωματικούς κανόνες και ρυθμίσεις. Όλα αυτά όμως διαγράφησαν λόγω τους ψήφους μας και γι' αυτό η ομάδα μου δεν θα μπορέσει να υπερψηφίσει την πρόταση αυτή. Λυπάμαι, λυπάμαι πάρα πολύ. Θα καταψηφίσουμε για τη συν Σίγουρα έχουμε ορισμένες βελτιώσεις και συμβαστικέ τροπολογίες, το μας πολύ σημαντικό το σημείο, είμαστε υποχρεωμένοι να καταψηφίσουμε, παραλαμβάνω. Okay. Well, I think, um, uh, Εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνω την απογοήτευσή σας. εκ μέρους όλων μας ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σκληρή δουλειά που κάνατε. Είναι μία γνωμοδότηση απλά, αλλά βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλο πολιτικό έργο από πίσω, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνατε. Ξέρω ότι πολλές φορές οι συγητές περιέρχονται σε δύσκολη θέση. Κυρία Κρόιτσφαλτ, θέλετε να πείτε κάτι. Και οι σκιώδεις συγητές έχουν το λόγο. Ε, καταρχήν θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά πόσο πολύ μου άρεσε η συνεργασία με την Κρίσταλ. Ίσως ε, κάποιοι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αναφώνησαν «Κοιτάξτε, καταρρύπτουν τις δικές τους ε, τροπολογίες». Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από το ΕΛΚΑ για την ενότητα που έδειξαν. Μερικοί συνάδελφοι ε, απέσυραν τις τροπολογίες τους, άλλοι τις καταψήφισαν και αυτό χάρη συμβιβασμού για να βρούμε μια λύση, για να συναντηθούμε στη μέση του δρόμου. Νομίζω ότι αυτή η ευελιξία θα πρέπει να ανταμυφθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους από το ΕΛΚ που το έκαναν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ας περάσουμε στην τελική ψηφοφορία γιατί πρέπει να εγκρίνουμε την γνωμοδότηση εν τέλει από την Επιτροπή μας. Περνάμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά με το ηλεκτρονικό σύστημα. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία. Να είστε πολύ προσεκτικοί παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την τελική ψήφο. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν 21 ψήφοι έναντι 15 ψήφων με 3 αποχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία με μια τόσο μακροσκελή ψηφοφορία και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως την εισηγήτρια αλλά και το προσωπικό μας που έκανε πολύ σκληρή δουλειά. Now we have a lot of other votes to do, so Πολλές ψηφοφορίες ακόμα, γι' αυτό σας παρακαλώ, όσοι εξέρχονται της αίθουσας, μήπως ήσυχα και ήρεμα μπορούν να εξέλθουν. Γιατί ακολουθεί κάτι το πολύ σημαντικό. Και, άλλες, και άλλα που θα πρέπει να ψηφίσουμε, έτσι. Το επόμενο σημείο λοιπόν είναι η έκθεση κυρία Χέντς.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 για την ψηφοφορία για την προστασία του καταναλωτή. Και έχουμε και πολλές τροπολογίες που κατατέθηκαν ε, πάνω από 80. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν από όλους. Ευχαριστώ τους συνεργάτες, τους συνεργάτες από την Επιτροπή επίσης και συμφωνώ με τον Σκιώδη Συγητή. Προσπαθήσαμε να πετύχουμε διάφορες, ε, να επικυρώσουμε διάφορες ε, συμβαστικές τροπολογίες, τροπολογίες ικανοποιητικές και ελπίζουμε και το αποτέλεσμα να είναι κάτι το καλό. Είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό και έχει σημασία να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για τον καταναλωτή. Ευχαριστώ. Θέλει εκ μέρους του ΕΛ και ο κύριος Μάρτιν επίσης να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια τη συνάδελφα Γιατί συμφωνώ ότι ήταν πολύ καλή η δουλειά, συνεργαστήκαμε πολύ καλά και όλοι συμφωνούν με το αποτέλεσμα. Εργαζόμαστε όλοι ώστε να έχουν περισσότερες δυνατότητες οι καταναλωτές πρόσβασης και χρήσης των δικαιωμάτων τους και είχαμε και μερικά σημεία πάνω στα οποία σκεφτήκαμε ότι χρειαζόταν να υποβάλουμε προτάσεις για να αποφύγουμε να προκύψει μία μη ισόρροπη έκθεση απέναντι σε όλους τους πολίτες που είναι και καταναλωτές αλλά και εργάζονται και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσοι παράγουν δηλαδή. Και θα πρέπει η εσωτερική αγορά να προσφέρει στους καταναλωτές τα δικαιώματά τους. Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε να αποφασίσουμε στη θέση των καταναλωτών. Μερικές φορές προσπαθώντας κάποιος να κάνει κάτι το καλό μπορεί να ξεπεράσει αυτή τη γραμμή και να είναι υπερβολικές οι κατευθυντήριες γραμμές και να ε, παγώσουμε αυτές τις παρεμβάσεις που δεν ευθυγραμμιζόταν με τα όσα έχουν να κάνουν με τη σημερινό πρόβλημα. Εντάξει, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει κανείς το τι γίνεται. Υπάρχουν πολλά μέσα, πολλά εργαλεία, θα πρέπει ήδη να ελέγξουμε τα όσα υπάρχουν ήδη και αν υπάρχει μια δραστηριότητα από πλευράς καταναλωτών να πληροφορηθούν για όσα μέσα τους προσφέρουν. Ε, υπόλοιποι. Εδώ ορισμένε προφορικές τροπολογίες. Είχαμε μικρό προβλήμα γραπτής μετάφρασης που άλλαξε όμως το νόημα δύο τροπολογιών. Εκεί που εμείς λέγαμε το public administration στα αγγλικά μπήκε σαν public authority Υπήρξε λοιπόν αυτή η διαφορά στη μετάφραση, έπρεπε να το διορθώσουμε στη γραπτή μετάφραση, διαφορετικά άλλαζε το νόημα και δεν θα είχε κανείς τη δυνατότητα ε, να εκφράσει κάτι το σωστά βασισμένο και αιτιολογημένο. Ευχαριστώ. Ουσιαστικά προτείνεται η προφορικές τροπολογίες αυτές να είναι επιπλέον ή υπάρχουν ήδη στο κατάλογο. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, να γίνει. Ε. Σίγουρα θα πρέπει να ζητήσω και τη σύμφωνη γνώμη. Δεν είναι στην κατάλογο ψηφοφορία, αλλά καθώ προχωράμε προτείνω να γίνει. Εντάξει, κατάλαβα. Θα πρέπει όμως, όπως ξέρετε, να γίνει προηγουμένως δεκτή από τον εισηγητή. Μόνο έτσι μπορεί να υποβληθούν την ημέρα της ψηφοφορίας προφορικές τροπολογίες. Περνάμε στην παράγραφο 1. 16 του κυρίου Τριανταφυλλίδη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 17 Ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. 18. Ροσφόρ. Υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Νομίζω ότι έχουμε ξεπράσει τον αριθμό αυτών που μπορούν να ψηφίσουν. Ποιος ψήφισε. Πρέπει να ελέγξουμε. Υπάρχει ένας επιπλέον. Φιλελεύθεροι. Πέντε φιλελεύθεροι. Τέσσερις. Υπάρχουν πολλοί φιλελεύθεροι, δεν ψήφισαν όμως όλοι. Υπάρχει ένας επιπλέον που ψήφισε. Ξαναψηφίζουμε λοιπόν. Ακυρώνεται η προηγούμενη ψηφοφορία και ξανά ψηφίζουμε. 39 είμαστε. 39 ψηφίζουν. Μάλλον 39 είναι παρόντες, 36 μόνο ψηφίζουν. 38. Τέλος ψηφοφορίας. 20 υπέρ 18 κατά. Εγκρίνεται. Η 19 καταπίπτει. 20 τριανταφυλλίδες υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. 39 παροντε τελος Τέλος. Εγκρίνεται. 19-18. Παράγραφος 4, Ιβάνοβα 21. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 5, Μότι και Κόμι. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 23, Τριανταφυλλίδης. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 24, Κάφα υπέρ, κατά, α, εγκρίνεται, συγγνώμη. Απορρίπτεται. Δεν θα έπρεπε να είχαμε ψηφίσει το 24, μου λένε. Γιατί αφού υιοθετήσαμε το 22, καταπίπτει. Παράγραφος 6, 25, μότι κόμι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 26, καταπίπτει. 27. Είναι προσθήκη της κυρίας Ιβάνοβα, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστικές τροπολογίες. Ένα παράγραφος 7. Ψηφίζουμε με ξεχωριστή ψηφοφορία. Βλέπετε τα τμήματα. Τμήμα 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το τμήμα 2 της συμβιβαστικής. Τέλος. Εγκρίνεται. 3. Τμήμα 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για το 4. Υπέρ. Μάλλον αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. 5. Ηλεκτρονικά ελέγχουμε. Δεν ξέρω τι ψηφίζει το ΕΛΚ. Τέλος. 33-3. Πέρασαν λοιπόν όλα τα κομμάτια. Ωραία. Ψηφίσαμε τμηματικά σε μια συμβιβαστική, αυτό είναι σπάνιο. Πέρασε λοιπόν η συμβιβαστική, άρα πάμε κατευθείαν στη 32. Πάκης. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7β καινούριο, 33. Υπέρ. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. 33. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 18 υπέρ 20 κατά. 34. 30 φιλίδης. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 8. Τροπολογία 35. Μότι και κόμι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8. Καινούριο. Τουν Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πρόκειται για την τροπολογία 36, 8α, 8 καινούριο. Τέλος. Απορρίπτεται. 17 υπέρ, 19 κατά. 9. Τροπολογία 17, μότι κόμι. 37, συγγνώμη. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Μότι και κόμι. Υπέρ. Α, χρειάζεται να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Και αναφέρομαι στην τροπολογία 39. 39. Αλλάζεται. Ψηφίζουμε για το 39. Τέλος. Εγκρίνεται 34-4. Για να αποφασίσω ναι ή όχι θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, βλέπω τις ενδείξεις. Η κυρία Γκέπχαρτ είναι σαφέστατη. Εσείς από το ΕΛΚ είστε λίγο πιο διστακτικός. Μπορείτε να μου δείχνετε την πρόθεσή σας έτσι ώστε κύριε Σφάπ να αποφασίζω και να επιταχύνουμε και τη διαδικασία. Δείξτε μου με σαφήνεια τι θέλετε να κάνετε. 38 είναι προσθήκη υπέρ. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 20-18. Και τώρα περνάμε στην 40 του κυρίου Τριανταφυλλίδη. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 16 υπέρ 22 κατά. 11. 42, τροπολογία 42, μότι κόμι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε. 41 καταπίπτει. Και περνάμε στην συμβαστική 2 και εδώ σε τρία τμήματα. Τρία τμήματα το πρώτο τμήμα της συμβαστικής 2 υπέρ. Κατά. Ομόφωνα εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 19-17. Το τρίτο τμήμα. υπέρ, υπέρ του τρίτου. Κατά. Δεν υπάρχουν αποχές, εγκρίνεται λοιπόν. Υιοθετείται λοιπόν όλο το κείμενο της συμβαστικής τροπολογίας και περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 3. Οι άλλες καταπίπτουν για την παράγραφο 15 υπέρ της 3. Κατά. Κανείς δεν είναι κατά, δεν υπάρχουν αποχές, εγκρίνεται λοιπόν. Προχωρήσαμε και πάμε στην 51. Όλες μέχρι την 51 καταπίπτουν. 51 λοιπόν του κυρίου Κάμφλη. Ψηφίζουμε τροπολογία 51. Τέλος. 15 υπέρ, 20 κατά απορρίπτεται. Κρόιτσμαν, έχετε αποσύρει. 55 του κυρίου Τριανταφυλλίδη, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 19. Τροπολογία head. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ροσφόρ 56 είναι μια προσθήκη. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ο κύριος Πουπάκης, προσθήκη, 57, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 56 και 57 εγκρίνονται λοιπόν. Αποσύρω την 59 ήταν για να γίνει σαφέστερο, αλλά τελικά δεν γίνεται. Περνάμε λοιπόν στην 60 με ξεχωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα πρώτα ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της 60. Τέλος. Απορρίπτεται. 33 κατά 3 υπέρ. 61, τροπολογία 61 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 23, 62. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 62. Πολύ αργά. Έχω ήδη ξεκινήσει την ψηφοφορία. Τέλος. 31 υπέρ, 6 κατά. 63, head. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, 20 κατά. 65 Πουπάκης 27 είναι η παράγραφος ποιος είναι υπέρ κατά εγκρίνεται 66 του κυρίου Τριανταφυλλίδη υπέρ α καταπίπτει 67 του κυρίου Πουπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ομόφωνα 28, παράγραφος 28 της κυρίας Χέντ η τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 μότι και κόμι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29α είναι η παράγραφος. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης έχει υποβάλει μια τροπολογία σε τρία τμήματα. Θα ψηφίσουμε. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Κάποιοι είναι υπέρ. Απορρίπτεται. Παράγραφος 31, 71, η τροπολογία του κ. Κάμφλιν. Υπέρ. Ηλεκτρονικά ελέγχουμε την 71. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. 20 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται. 32 παράγραφος 32. Τροπολογία μότι κόμι 72. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 73 μάντελς Αποσύρω και αυτή την τροπολογία. Όλοι είναι κατά. Για μένα ήταν σημαντικό να μιλήσουμε για το επιπλέον διοικητικό άκθος. Την αποσύρω πάντως. Περνάμε στην 74, είναι δική μου, να την υποστηρίξετε λοιπόν. Ελπίζω το ΕΛΚ, ο κύριος Φαμπ δεν προσέχει. Ευχαριστώ. Ποιος είναι κατά της τροπολογίας μου? Είστε κατά. Χωρίς αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν η τροπολογία μου. 64 της κυρίας Χέντ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 75 του κυρίου Τριανταφυλλίδη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 76 Κρόιτσμαν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στην 80 Το κύριο Πουπάκη. Υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 80. Τέλος. εγκρίνεται 23 υπέρ 15 κατά 81 μότι και κόμι υπέρ κατά εγκρίνεται Ακούστε πρόεδρε Μήπως την προφορική τροπολογία για την 82 τροπολογία της παραγράφου αυτής, αυτό να κάνω και τι ζητάμε. Αντί για το public administration που αναφέρεται εκεί, που μπήκε κατά λάθο στη γραπτή μετάφραση το public authority, να βάλουμε τη φράση public and organizations providing services ε, για να καταλάβουν καλύτερα ότι μιλάμε για τις υπηρεσίες προσφέρονται στους καταναλωτές από νοσοκομεία είτε και κάπως λιγότερο για, για τις μεταφορές αλλά όχι από ιδιωτικές εταιρείες. Αν κατάλαβα καλά, έπρεπε αυτό να γίνει πριν ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο που μιλάει για αρχές, δημόσιες αρχές. Συμφωνείτε με το κείμενο που προτείνετε, κυρία Χέντ. Ναι, όχι. Ακούστε, ε, εντάξει, αν θέλετε να επιφέρετε την αλλαγή αυτή, μπορείτε να το κάνετε. Κανένα πρόβλημα. Uh, να ξαναδιαβάσουμε λοιπόν το κείμενο. Πρόεδρε, πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει κάτι να διευκρινίσουμε. σε ορισμένες μεταφράσεις ε, ή παραγράφους μάλλον ε, τροπολογίες να διορθώσω ακόμα λέει ο μιλητής. Εδώ ήταν μία αλλαγή αλλά μία ενσωμάτωση. Να σας το διαβάσω στα Ιταλικά όμως το έχω το κείμενο αυτό το άρθρο έτσι με αυτό που ενσωματώνω εγώ την τροπολογία αυτή στην οποία ενσωματώνω το μέρος αυτό. Θέλω να σας το διαβάσω. Προσθέτουμε δηλαδή εδώ, με αυτή την προφορική τροπολογία, το public authority, δημόσιες αρχές. Ναι, εκεί το ενσωματώνω που αναφερόταν μόνο οι διαφωνίες με επαγγελματίες και με τη δημόσια διοίκηση για να αποφύγουμε λάθος ε, που το λέμε public and organizations providing services. Έτσι το λέμε. Ε, ε, τα καταλαβαίνετε τι ζητάω τώρα εγώ σαν τροπολογία, με καταλαβαίνετε. Το είδαμε το πρόβλημα την τελευταία στιγμή και δεν καταλαβαίναμε γιατί δεν συμφωνούσαμε οι μεν με τους δε. Γιατί η μετάφραση δεν ήταν η σωστή ή καλή που να σέβεται το την πρωτότυπη τροπολογία. Μπερδευόμαστε λοιπόν. Άρα θα αντικαταστήσουμε αυτήν την φράση, αυτό το κομμάτι και ψηφίζουμε. Θέλετε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. 83, Κρόιτσμαν. Και τώρα περνάμε στην παράγραφο 40. 83, τροπολογία 83, Κρόιτσμαν. Ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά, τροπολογία 83. Τέλος. 18-18. Απορρίπτεται. 84. Ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 44, παράγραφος 44, υπάρχει μια προφορική τροπολογία, πρέπει να την έχετε στον κατάλογο, γραπτά, είναι της εισηγήτριας και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. 22 υπέρ, 14 κατά. Τροπολογία 85 καταπίπτει. 86 Κρόιτσμαν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 87 Κρόιτσμαν. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Ψηφίζουμε την τροπολογία της κυρίας Τούρμ. Τροπολογία 1. Τέλος. Απορρίπτεται 18 υπέρ 19 κατά. 2. Δική μου τροπολογία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 2. Ψηφίζουμε. Πολύ πολύ αργά ψηφίζεται σήμερα. Τέλος. Εγκρίνεται. 19-16. 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4. Μότι κόμι υπέρ. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. 4. Για την 4 ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 14 υπέρ 23 κατά. 5. Τροπολογία 5. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 5. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 19 υπέρ 18 κατά. 6, τροπολογία 6 του κύριου Μότη και της Κόμη. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, 23 κατά. Τροπολογία 7. Υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8 του 30 Τριανταφυλλίδη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 9 κύριο 30 Τριανταφυλλίδη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 10 κυριο 30 Τριανταφυλλίδη. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Απορρίπτεται. 15 υπέρ 22 κατά. 11 του κυρίου Μότη. της Σκόμη Έχω τη δεύτερη προφορική τροπολογία πάνω σε αυτό. Έτσι. Ναι, προχωρήστε. Πέστε μας. Ναι, να σας πω ότι έχουμε και από τη Δημοσιοδιοίκηση υπηρεσία και να διαβάσω τη σύντομη τροπολογία ακριβώς να τη υπόψη ότι θα πρέπει οι κατανοητέ να μπορούν ε, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους όταν είναι θύματα παράνομων ενεργειών είτε από ιδιωτικό τομέα είτε από public ε, και λοιπά provided services που είναι ουσιαστικά το δημόσιο. Εντάξει, για να αποφύγουμε τον λαθασμένο όρο που είπαμε πριν στα αγγλικά. Ζητάτε ουσιαστικά την ίδια ακριβώς διατύπωση. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 11. Τέλος. Απορρίπτεται. 17 υπέρ, 20 κατά. 12, τροπολογία 12. Ψηφίζουμε την τροπολογία 12. Τέλος. 19 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται. Του κυρίου Τριανταφυλλίδη είναι η επόμενη τροπολογία. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 22 υπέρ, 15 κατά. Προφορική 40 της κυρίας Χέτ. Την έχετε στο κείμενό σας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 14 καταπίπτει νομίζω. Η τελική είναι η 15 της κυρίας Ιβάνοβα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το τελικό κείμενο. Κυρία Χέτη, είστε ευτυχείς. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας για το κείμενο της έκθεσης. Τέλος. 34 υπέρ, καμία ψήφος κατά, τρεις αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Χέτ. Συγχαρητήρια. Και σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Άρα δεν υπευλήθησαν οι τροπολογίες με τον παραδοσιακό τρόπο. Και ελπίζω στην Ολομέλεια να έχουμε εξίσου ενδεικτική ψηφοφορία. Η μία... Έχουμε δύο κείμενα να ψηφίσουμε για τον κύριο Τύρμε. Συγγνώμη κύριε Τούρμε που σας κάναμε να περιμένετε. Έχετε να πείτε κάτι πριν περάσουμε στην ψηφοφορία των δύο κειμένων σας. Θέλω απλώς να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, την κυρία Παβανόβα, την κυρία Βερνιού, τον κύριο Ζουβέρ, τον κύριο Φόξ από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Νομίζω ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά και ότι θα είμαστε ικανοί να ψηφίσουμε και πολλές συμβιβαστικέ τροπολογίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το δικό του προσωπικό, το δικό μου προσωπικό και να σας συγχαρώ ε, κύριε Πρόεδρε για το εξαιρετικό έργο της Γραμματείας. Πραγματικά η Γραμματεία μας βοήθησε πάρα πολύ να φτάσουμε εδώ που ήρθαμε. Αυτά ήταν όλα που είχα να πω. Uh, ε, να σας θυμίσουμε ότι καταρχήν στην αρχή θα ψηφίσουμε την οδηγία. Άρθρο 11 της οδηγίας υπάρχει μια ενοποιημένη τροπολογία από τους σοσιαλιστές, τους δημοκράτες, τους πράσινους και την ECR. Ποιοι είναι υπέρ, νομίζω κατευθείαν θα ξεκινήσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία για την τροπολογία 1. The vote is closed. Oh, we've got 40 votes take it again. All right, sorry. There were 16, 16. Uh, sorry, we had, we had more people voting. So... Συγγνώμη, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που ψηφίζουν, επομένως ε, μάλλον έχουμε περισσότερους να ψηφίζουν από αυτούς που πρέπει να ψηφίζουν. Αυτό έλεγα, ότι είναι πολλοί αυτοί που ψηφίζουν και το σύστημα δεν μας επιτρέπει να δούμε από ποια πολιτική ομάδα προέρχονται. Παρακαλώ μπορείτε να ελέγξετε τους αριθμούς σας. There 40, άτομα δικαιούνται να ψηφίσουν. Κάποιες πολιτικές ομάδες έχουν φέρει παραπάνω. Νομίζω ότι είμαι 41 ότι ψήφισαν. Πρέπει να το ελέγξουμε. Μπορούμε να περατώσουμε αυτή την ψηφοφορία. Παρακαλώ να δούμε ποια μέλη του ΕΛΚ ψήφισαν ευνοϊκά, ψήφισαν θετικά. 15 είναι ένας ο ένας πλεονάζει. 14. Οκ. Εντάξει. Ωραία. Ας δούμε την ψηφοφορία μας τώρα. Ενοποιημένη τροπολογία 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 19 έναντι 18. Καλά κάναμε λοιπόν και ελέγξαμε τους αριθμούς. Αυτό σημαίνει ότι τώρα θα περάσουμε στην τροπολογία 35 της κυρίας Φόξ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Κλοντ Τούρμς έχουν αποσύρει την 6. Είμαστε στην 36 από αρκετούς διακεκριμένους βουλευτές. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 37 της κυρίας Φερνιό. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 38 της κυρίας Βερνιό. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Άρθρο 27. Τροπολογία 39 της κυρίας Βερνιό. Υπέρ, κατά, Μπορούμε να το ελέγξουμε παρακαλώ. Τροπολογία 39 της κυρίας Βερνιό. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 23 κατά, 15 υπέρ. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της τροπολογίας Βερνιό. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 15 υπέρ 38 κατά. Τροπολογία 41 του κυρίου Ζουβά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 42, 43, 44, 45, όλες τις κυρίες βερνιωθη θα τις ψηφίσουμε unblock, όλες μαζί. Αρχίζει η ψηφοφορία για τις τέσσερις αυτές τροπολογίες. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτονται 15 υπέρ 38 κατά. Τροπολογία 46 της κυρίας Βερνιό. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Οι 7 καταπίπτει λοιπόν. Άρθρο 59. Αυτές οι τροπολογίες καταπίπτουν γιατί η ενοποιημένη τροπολογία εγκρίθηκε Τώρα τι γίνεται με το 46, με, το με τη 48. Οι 48 και 49 καταπίπτουν και αυτές. Όχι. My Ο Κλοντ Τούρμα. Σχετικά προς το τέλος της ψηφοφορίας θα ψηφίσουμε την τροπολογία 3 και θα πρέπει τότε να επανέλθουμε να ψηφίσουμε την 48 και 49. Η τροπολογία 3 είναι στην τελευταία σελίδα του δικού μου κειμένου τουλάχιστον. Μα πρώτα ψηφίζουμε τα άρθρα και μετά τις αιτιολογικές σκέψεις. Οι αιτιολογικές σκέψεις δεν έχουν το ίδιο νομικό βάρος με τα άρθρα. Οπότε δεν είμαι βέβαιος ε, πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Μου φαίνεται λίγο αλόκοτο Νομίζω ότι καλύτερα είναι να ψηφίσουμε τώρα αυτές τις τροπολογίες. Λοιπόν, 48. Αρχίζει η ψηφοφορία. Είναι της κυρίας Παρβανόβα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 49 της κυρίας Βάισγκαρμπερ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 49. Πέρα τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 37 κατά, 14 υπέρ. Περνούμε τώρα στην τροπολογία 51 για το άρθρο 65. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50, το πρώτο τμήμα της κυρίας Παρβανόβα. Νομίζω ότι αυτό καταπίπτει. Μ, ναι. Το δεύτερο μέρος. Μπορούμε να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 50. Το δεύτερο τμήμα. Το πρώτο καταπίπτει. Ποιοι είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. 50, δεύτερο τμήμα. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 συν μία αποχή. Τώρα 10 του κυρίου τύρμη για το άρθρο 102, χωριστή ψηφοφορία μετά από αίτηση του ΕΛΚ. Θέτω το πρώτο τμήμα σε ψηφοφορία. Κατά ε, εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Απορρίπτει. κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 22 σύν, 14 κατά και 2 αποχές. Η 52 καταπίπτει. Η τροπολογία 11 του κυρίου Τούρμε. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 του κυρίου Τούρμε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53 της κυρίας Βερνιού. Υπέρ. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 53. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ, 22 κατά. Περνούμε στην ενοποιημένη τροπολογία 2. Από τους σοσιαλιστές δημοκράτες και τους πράσινους. Κλοντ. Ναι. Εδώ έχουμε μια προφορική τροπολογία. Αυτή η προφορική τροπολογία έχει μοιραστεί σε όλους σας. Θα πρέπει... Θέλετε παρόλα αυτά να τη διαβάσω. Όχι, νομίζω ότι όλοι την είδαν. Και αν την δέχεται η Επιτροπή να ψηφίσει επί της τροπολογίας αυτής, εντάξει. Δεν ξέρω ποια είναι η πρόθεση σας. Ωραία, θα ψηφίσουμε την ε, ενοποιημένη τροπολογία 2 όπως τροποποιήθηκε με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει... Η... Α, η 13 Αποσύρθηκε η 54 καταπίπτει. Περνούμε στο άρθρο 106, τροπολογίες 55 και 56. Αρχίζει η ψηφοφορία. Κατά. Κλείνει η ψηφοφορία. 19-19, επομένως απορρίπτεται. Οι 55 και 58 καταπίπτουν γιατί ψηφίσαμε την ε, ενοποιημένη τροπολογία 1. Ε, τροπολογία 14 του κ. του υπέρ, υπέρ της 14, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογίες 59 και 61. Είναι χωριστή ψηφοφορία. Έχουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα. Το πρώτο τμήμα της 61, ας το πούμε έτσι. Είναι ταυτόσιμες οι δύο τροπολογίες. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της, κυρίας, της τροπολογίας αυτής, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Επομένως καταπίπτουν τώρα οι τροπολογίες του κυρίου Φόξ και έχουμε μια άλλη τροπολογία του κυρίου Φόξ, την 62. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Άρθρο 107, τροπολογία 63 του κυρίου Ζουβά, υπέρ, κατά, απο, εγκρίνεται. 64 του κυρίου Ζουβέν υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Επομένως καταπίπτουν οι 15, 16 και 65. Τροπολογία 17. Ποιοι είναι υπέρ. Μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 17 υπέρ, 19 κατά. Ε, συγγνώμη, 19 κατά, 17 υπέρ και μία αποχή. 18 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 66 του κυρίου Ζουβέν υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα, περνάμε στην ε, 19 του κυρίου Κλώτου Τούρμε, το πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 68 του κυρίου Ζουβέν, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 69 του κυρίου Ζουβέν, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 20 του κυρίου Τούρμ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα, 21. Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα της 21. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 20 υπέρ, 16 κατά μία αποχή. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 70 της κυρίας Παρβανόβα. Υπέρ. Κατά. Νομίζω πρέπει να το ελέγξουμε. Μπορούμε παρακαλώ. Της κυρίας Παρβανόβα η τροπολογία 70. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 27 συν 11 κατά. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Επομένως η 71 του κυρίου Ζουβέν καταπίπτει. Σε 72 του κυρίου Ζουβέν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 22 του κυρίου Τούρμ υπέρ. Κατά. Μπορούμε να το ελέγξουμε παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 22. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 15 υπέρ 22 κατά μία αποχή. Άρθρο 2. Τροπολογία 73 του κυρίου Ζουβέν. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 74 της κυρίας Ράπτη. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 22 της κυρίας Παρβανόβα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. λογική σκέψη 9, τροπολογία 24 της κυρίας Παρβανόβα. Τώρα. Ας ψηφίσουμε ούτως ή άλλως. 24 της κυρίας Παρβανόβα. Α. Όχι, καταπίπτει, όπως και 25. Οπότε δεν ψηφίζουμε για αυτές. Περνούμε στην τροπολογία 26.1 ε, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και τροπολογία 2, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 της κυρίας Βερνιό, υπέρ, Α, αποσύρει η κυρία βερνιό την 27. Περνούμε στην 28 του κυρίου Ζουβέν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αντιλογική σκέψη 17, τροπολογία 29 της κυρίας Βεγνιό. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 29. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 24 κατά, 15 υπέρ. Τροπολογία 3 του κυρίου Τύρμες. Υπέρ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 29 υπέρ, 20 υπέρ, 18 κατά μια αποχή. 20, 30 του κυρίου Ζουβέν υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 31 της κυρίας Βερνιό. Α, την αποσύρει, μάλιστα. Περνούμε στην τελική ψηφοφορία τότε. Η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 38 υπέρ, κανένας, καμία ψήφος κατά, μία αποχή. Κύριε Τούρμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και περνούμε τώρα στον κανονισμό. Πάλι είναι εισηγητής ο κύριος Τύρμ. Κλοντ, θες να πεις, κα... θες να πεις κάτι? Στην σελίδα 5, για την 67, δεν την είχαμε, αλλά επειδή έχει διανεμηθεί μπορούμε να συνεχίσουμε. Ας περάσουμε στον κανονισμό λοιπόν τροπολογία 13 της κυρίας Βερνιό έχει αποσυρθεί. Περνάμε στην τροπολογία του κυρίου Ζουβέν 12. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 14 της κυρίας Βάισπικερμπερ. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 1 του κυρίου Τύρμα. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 του κυρίου Τύρμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 της κυρίας Βερνιό. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 του κυρίου Τύρμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 του κυρίου Φόξ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 16. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24 ψήφοι υπέρ, 15 κατά, καμία αποχή. Τροπολογίες 17-18, Fox και Βάις υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Τροπολογίες 19 και 20, Fox και Γκέρμπερ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21, και 22. Vice Gerber Fox, ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 21, το δεύτερο μέρος της κυρίας Vice Gerber, υπέρ. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 21, το δεύτερο τμήμα, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίες. ψηφοφορια Εγκρίνεται 28 συν 19 κατά μία αποχή. Η 23 καταπίπτει λοιπόν κατά αποτέλεσμα. Η 24 της κυρίας Παρβανόβα. Υπέρ. Θα κάνετε προφορική τροπολογία. Παρακαλώ. Η πρώτη, το πρώτο τμήμα... Προτείνω να διαγραφεί αυτό το κομμάτι και το υπόλοιπο κείμενο να μείνει ως έχει. Νομίζω ότι την έχετε διανύμει, την λάβατε όλοι. Ποιο είναι υπέρ του κειμένου όπω τροποποιήθηκε από την κυρία Παρβανόβα. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην 25 του κυρίου Φόξ, άρθρο 27. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 26 της κυρίας Βερνιό, αρχίζει η διαδικασία Αρχίζει η ψηφοφορία για την 26. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 15 υπέρ 24 κατά. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Ενοποιημένη τροπολογία. Η συμβιβαστική τροπολογία και πάλι έχετε το κείμενο, το διένυμε ο κύριος Τούρμα. Α, όχι, συγγνώμη, αυτή ήταν η συμβιβαστική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται. Επομένως, 27 καταπίπτει. Τροπολογία 28 της κυρίας Βερνιό. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 του κυρίου Τούρμα, νομίζω καταπίπτει. Τροπολογία 29 της κυρίας Βερνιό. Α, την απέσυρε, μάλιστα. Περνούμε λοιπόν στην τροπολογία 30 της κυρίας Βερνιό. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 30. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14 υπέρ 22 κατά. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Λοιπόν. η 31 καταπίπτει. Έχουμε τις 32, 33 και 34. Τις αποσύρετε. Α, ναι, αποσύρθηκαν αυτές. Την 35 θα την ψηφίσουμε, κυρία Βερνιό. Ναι. Υπέρ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 14 υπέρ, 23 κατά. Τώρα, τροπολογία 5 του κυρίου Τύρμ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ενοποιημένη τροπολογία 1 με το κείμενο που είναι η προφορική τροπολογία που αναφέρατε. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι περνούμε στο άρθρο 2, τροπολογία 7 και 37. Τον Τουρμ και Ζιβέν. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η τροπολογία 38 της κυρίας Παρβανόβα καταπίπτει. Τροπολογία 9 της κυρίας Βερνιό. Α, αποσύρθηκε. Εντάξει. Τροπολογία 8 του κυρίου Ζουβέν, λοιπόν. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 10 της κυρίας Βερνιό. Α, καταπίπτει νομίζω. Α, αποσύρθηκε. Εντάξει. Η 10 αποσύρθηκε. Νομίζω είχαμε ήδη ψηφίσει την 26. Η τροπολογία 11 της κυρίας Βάις Γκέρμπερ. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία λοιπόν, ηλεκτρονικά. Ψηφοφορία για την ε, γνωμοδότηση. Άρχισε η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 37 υπέρ καμία κατά και μία αποχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κλοντ Τύρμα. Νομίζω ότι σου αξίζουν κάποια χειροκροτήματα. Είναι πολύ ωραία να κάνει κανείς πιο πολλές ονομοδοτήσεις παρά εκθέσεις. Είσαστε πάντοτε ευπρόσδεκτος στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Ναι, νομίζω πρέπει να τα δούμε και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος αυτά. Τώρα θα περάσουμε στις δύο τελικές γνωμοδοτήσεις της ε, κυρίου Μπουζόη, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Όσοι θα φύγετε μετά την φαρμακοεπαγρύπνηση, μπορείτε να το κάνετε παρακαλώ ήσυχα για να μπορέσουμε εμείς να συνεχίσουμε. Κύριε Μπουζόη, θέλετε να λάβετε το λόγο. Χαίρομαι πάρα πολύ που η πρώτη μου έκθεση τράβηξε το ενδιαφέρον τόσων συναδέλφων. Έχουμε τόσες πολλές τροπολογίες, συμφωνώ με τις περισσότερες. Νομίζω ότι αυτή η συνεισφορά κάνει πολύ θετική την έκθεση. Ε, σας προτείνω να υπερψηφίσετε αυτήν την γνωμοδότηση και Έχω και μια προφορική ε, τροπολογία να κάνω κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, την οποία συμφώνησα με όλες τις πολιτικές μου ομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ στους παρεμβαίνοντες, τους σκιώδεις εισηγητές και το προσωπικό, καθώς και τη γραμματεία. Πρόεδρος, οκ, okay, ας ξεκινήσουμε. Γιατί έχουμε πολλές ψηφοφορίες, δεν θέλω να καθυστερούμε. Περνούμε λοιπόν στην ψήφιση της έκθεσης του κυρίου Μπουζόη. Τροπολογία 8 της κυρίας Ρόιτοβα και του κυρίου Πουπάκη. Ποιοι είναι υπέρ κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ρόιτοβα και Χόχενστάιν. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Κύριε Γκρέχ, υπέρ του κύριου Γκρέχ. Εγκρίνεται. 11. Του Ντεγιόνγκ και άλλων. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τη κυρία Ρόιτοβα, 13. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τη κυρία Στίλερ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται του κυρίου Γκρέχ. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δε Γιόγκ και άλλων, 12 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Του κυρίου Μπουζουτήλ από την Επιτροπή Αναφορών υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 6, τροπολογία 16 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Από την Επιτροπή Αναφορών του κυρίου Μπουζουτήλ υπέρ, καλά, Κατά. Ε, εγκρίνεται. Της κυρίας Ρόιτοβα η 17 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Ρόιτοβα και Πουπάκης υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Της κυρίας Στάιλ Η 20 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 21 της κυρίας Ρόιτοβα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 22 της κυρίας Στήλερ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα, συμβιβαστική τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ της συμβιβαστικής τροπολογίας 1, κατά, εγκρίνεται. Επομένως, ε, περνάμε τώρα κατευθείαν στην τροπολογία 29. 29, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα έχουμε όλες αυτές τις τροπολογίες από την Επιτροπή Αναφορών. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Λοιπόν, προτείνω όλες τις τροπολογίες της Επιτροπής Αναφορών από την 3 μέχρι την 11, 12, να τις ψηφίσουμε από κοινού υπέρ, κατά, εγκρίνονται όλες. Συμβιβαστική τροπολογία 2, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 31 του κυρίου Λόκεγκάρντ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12, τροπολογία 32, ντεγιόν και άλλων. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 33 του κυρίου Γκρέκ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 35 της κυρίας Στίλερ. Ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 34 του κυρίου Μπουζόη ως προσθήκη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 37 της κυρίας Ροϊτοβά υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και 36-37 καταπίπτουν. 38 και 36 καταπίπτουν. Περνάμε στην 39. Μπορούμε να ψηφίσουμε όλες μαζί τις τροπολογίες της κυρίας Ρόιτοβα. Ναι. Όλες λοιπόν 39, 40, 41, 42, 43, όλες μαζί, υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Τροπολογία 44, Κρόιτσμαν, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και 45 του κύριου Κάρας, ως προσθήκη, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα, τη λογικές σκέψεις, ε, τροπολογία 1 του κύριου Κρόιτσμαν, μπορούμε και όλες μαζί, προτείνει ο εισηγητής όλες τις τροπολογίες των αιτιολογικών σκέψεων. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνονται και πρέπει ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε και την έκθεση εν συνόλο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Μπορώ και εγώ να ψηφίσω. Δικαιούμαι και εγώ. Ψηφίζω και εγώ για να δείξω την αλληλεγγύη μου. Ψηφίζω υπέρ. Ωραία, πέρα ψηφοφορία, τρόπο ψήφισα κι εγώ. 34 υπέρ, 2 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για την πρώτη και πολύ επιτυχή σας έκθεση. Και τέλος ψηφίζουμε στην uh, τελευταία έκθεση Θέλετε να πάρετε το λόγο. Όπως είπε ο κύριος Τούρμες, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ενασχόληση το να παρουσιάζει κανείς τέτοιες εκθέσεις πρωτοβουλίας, νομοδοτήσεις πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Τερέζα Πίντο και τους σκιώδεις γιατί πραγματικά με βοήθησαν να, να βελτιώσω το κείμενο. Ευχαριστώ λοιπόν τους ε, Σκιώδης. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε λοιπόν. Παράγραφος 1, τροπολογία Κέλλη, εγκρίνεται. 3, τροπολογία 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τουν Κέλλη, τροπολογία 4 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 6. Πουπάκης υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τε Ιόγκ είναι προσθήκη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τουν και Κέλλη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ρόιτοβα, έχει αποσυρθεί. Τε Ιόγκ Νομίζω πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 9. Τέλος. 15 υπέρ 20 κατά. Απορρίπτεται. Ο κύριος Πουπάκης. Δεκατρία υπέρ κατά εγκρίνεται. Κυρία Ρόιτοβα, έχει αποσυρθεί. Όχι, α, καταπίπτει. 11. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, γιατί η τροπολογία 11. Τέλος. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, 24 κατά. Ε, συμβιβαστική τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Καταπίπτουν κάποιες τροπολογίες. Συμβιβαστική 2. Ποιος είναι υπέρ. Τα. Εγκρίνεται. 21. Σαν προσθήκη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 22. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά εγκρίνεται. 26. Νομίζω πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 26. Ψηφίζουμε για την 26. Τέλος. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, 24 κατά. 27 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. λογικές σκέψεις. Τροπολογία 1. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίνουμε τώρα όλο το κείμενο της γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. 13, ε, συγγνώμη, 32 υπέρ, μία ψήφος κατά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλους τους ε, εισηγητές, όλους εσάς. Κράτησε πολύ αυτή η ψηφοφορία, αλλά τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Επειδή η ψηφοφορία κράτησε πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι είχαμε προβλέψει, ο χρόνος μας πιέζει. Υπάρχουν διάφορα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Γι' αυτό και θα ήθελα να πω στους συντονιστές ότι θα έχουν μόνο μισή ώρα για να δώσουμε μισή ώρα στην κυρία Βάλα. Συμφωνείτε? εντάξει, για τις ε, καθημερι... καθυστερημένες πληρωμές. Μισή ώρα έχετε. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ καθίστε. Η αίθουσα είναι μικρή. Κύριε Βάλερ, έχετε μισή ώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους συντονιστές που μπορούμε έτσι άτυπα να πάρουμε αυτή την απόφαση. Μισή ώρα φτάνει, μισή ώρα φτάνει, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και τις τροπολογίες έτσι ώστε όλες οι πολιτικές ομάδες να μπορέσουν από την επόμενη εβδομάδα να υποβάλουν τροπολογίες. Οι περισσότεροι που έχουν παρακολουθήσει το θέμα αυτό ξεκινήσαμε τη συζήτηση τον Νοέμβριο γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται και γνωρίζουν ότι οι τροπολογίες ε, θα ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Θα επικεντρωθώ στα πιο σημαντικά σημεία μόνο. Πρώτον, έγιναν όπως ξέρετε συζητήσεις και ακροάσεις με εμπειρογνώμονες αλλά και με μέλη των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων Συζητήσαμε επίσης με τους εκπροσώπους των διαφόρων φορέων σε εθνικό επίπεδο και το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων είναι ότι και στον ιδιωτικό και στον ε, δημόσιο τομέα θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να καθοριστούν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις χωρίς, ε, αν θέλετε, να ξεκινήσει η διαδικασία της ε, διαφοράς της αντιπαραβολής. 5% αν θέλετε αυτών των ε, υποθέσεων φτάνουν τελικά στο δικαστικό τομέα. Εγώ θέλησα καταρχήν να ξαναδώ όλες τις ε, προθεσμίες. 30 ημέρες είναι στις περισσότερες ε, χώρες η αρχική προθεσμία, αλλά θεωρώ ότι περίπου 1%, 0,5% είναι τελικά το ποσοστό των υποθέσεων που παρόλα αυτά και μερά, μετά από αυτήν την προθεσμία των 30 ημερών, συνεχίζουν και μπαίνουν στη διαδικασία των εκκρεμών υποθέσεων. Θα ήθελα επίσης εδώ να σας πω ότι οι διάφοροι τομείς που μας απασχόλησαν και που εξετάσαμε και εδώ αναφέρομαι στο άρθρο 17, στην οδηγία 17 και 18. Όπως ξέρετε υπάρχουν διάφορες ε, οδηγίες στις οποίες μπορούμε να αναφερθούμε, αλλά ιδιαίτερα στο άρθρο 17, στο άρθρο αυτό, η ερμηνεία μου είναι ακριβώς αυτή που όλοι θέλατε, αυτή που όλοι περιμένετε, να υπάρχουν ίδιοι κανόνες και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουμε ζητήσει από την Επιτροπή όχι μόνο δηλαδή αιτιολογική σκέψη, αλλά άρθρο στο κείμενο και ελπίζω να με στηρίξετε στην Ολομέλεια εάν αυτό είναι κάτι που τελικά αμφισβητηθεί. Τώρα, όσον αφορά τους ε, τόκους ε, υπερημερίας, η Επιτροπή κάνει κάποιες προτάσεις και προτείνει εδώ ένα ποσό 10.000 ευρώ, 1% το θεωρώ ίσως υπερβολικό εδώ. Κάνω μια άλλη πρόταση και μιλάω για ένα συνολικό ποσό 100 ευρώ. Προσπάθησα να βρω έναν τρόπο να γίνει η συμπερίληψη αυτών των προτάξεων είτε παραδείγματο χάνει για ό,τι έχει σχέση με το δημόσιο τομέα, για τα νοσοκομεία, παραδείγματο χάνει τα κρατικά. Ζητούμε περισσότερη ευελιξία. 60 μέρες είναι η πρώτη πρόταση με μία μοναδική εξαίρεση. Αλλιώς για όλες τις άλλες περιπτώσεις παραμένουμε στις 30 ημέρες. Εκτός από κάποιες ειδικέ εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούμε να δεχτούμε τις 60 ημέρες. Για τα νοσοκομεία 60 μέρες νομίζω είναι κάτι που μπορούμε να το δεχτούμε στη Γερμανία παραδείγματος και σε άλλες χώρες υπάρχουν πάρα πολλά νοσοκομεία που καταβάλουν τις πληρωμές τους Εγκέρος, Άλλες περιπτώσεις μας δείχνουν ότι η κατάσταση σε κάποια νοσοκομεία είναι εξαιρετικά δυσάρεστη. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει οι μεν να ενημερωθούν ε, και να μάθουν από τους δε. Προσπάθησα να μεταφράσω κάποιες αγγλοσαξονικές έννοιες, γιατί εμπνευστήκαμε από το βρετανικό σύστημα. Μπορούμε να μιλήσουμε εδώ για κυρώσεις, για ένα άγριο ζώο το οποίο φοβάται κανείς, αλλά το οποίο τελικά δεν είναι τόσο τρομερό. Πρέπει δηλαδή να δούμε την θετική επίδραση αυτού του συστήματος την αποτροπή αν θέλετε πριν φτάσουμε στις ε, κυρώσεις. Πιστεύω όμως ότι τα κράτη-μέλη, αν και δεν είναι υποχρεωμένα να υιοθετήσουν αυτή τη σειρά μέτρων, θα μπορούσαν να το κάνουν. Αυτά είναι τα σημεία που θα ήθελα να σας παρουσιάσω. Βεβαίως υπάρχουν εδώ πάρα πολλές ε, επικρίσεις που μας υπέβαλαν, παράδειγμα του χάρη, οι δημικοί κοινότητες. Είχα το πάρα πολύ δύσκολο φαινόμενο αυτών που δεν ήθελαν καθόλου να ρυθμιστεί ο τομέας. Άλλοι που ήθελαν να γίνει πολύ πιο αυστηρό το κείμενο και να συμπεριληφθούν κι άλλοι τομείς, όπως αυτών των καταναλωτών παραδείγματος χάρη. Βρήκα λοιπόν μια μέση λύση. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν έλαβα υπόψη μου τις πολύ αυστηρές κριτικές των κοινοτήτων από τη μία, αλλά και την ε, πολύ αυστηρή πρόταση της Επιτροπής από την άλλη, όσον αφορά τις καθιστεμένες πληρωμές. Επίσης έχουμε και την πρόταση της ε, Επιτροπής Νομικών ε, Υποθέσεων, έχουμε και τις τροπολογίες. Το ερώτημα είναι αν αυτή η οδηγία θα είναι μια βελτιωμένη έκδοση της οδηγίας του 2000. Και βεβαίως Ελπίζω οι τροπολογίες που τελικά θα υιοθετηθούν θα έχουν σαν αποτέλεσμα να βελτιωθεί η κατάσταση, να βελτιωθεί η ρευστότητα και να υπάρξουν καλύτερες δυνατότητες και καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Σφάμπε, θέλετε να πάρετε το λόγο εκ μέρους του ΕΛΚ. Ο κύριος Κρότσμαν είναι εδώ, η κυρία Ρούλε. Ο κύριος Ντεγιόγκ όμως έφυγε. Σύντομες παρατηρήσεις, μην ξεχνάτε το χρόνο. Έχουμε και το Συμβούλιο εδώ. Η κυρία Μπρίκμαν είναι εδώ εκ μέρους της Επιτροπής. Εάν μας μείνει λίγος χρόνος θα σας δώσω το λόγο. Ας ξεκινήσουμε όμως με τον κύριο Σφάμπα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν εξ ονόματος της α, εισηγήτριας, της σκιώδους εισηγήτριας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βέλλα για την εξαιρετική συνεργασία. Δεν είναι σήμερα παρούσα η σκιώδης εισηγήτρια, αλλά μου ζήτησε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν είναι πολύ σωστή η πρόταση της κυρίας Βέλλερ. Στα περισσότερα ε, σημεία συμφωνήσαμε, κάποια τα ενδυναμώσαμε και κάποια προσπαθήσαμε να τα αποδυναμώσουμε. Αλλά η βασική ιδέα είναι η ίση μεταχείριση όλων των φορέων της αγοράς. Είναι δύσκολο πολλές φορές κάποιος να κάνει διαχωρισμό μεταξύ φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Σκοπός μας είναι πάντως να υπάρξει ίση μεταχείριση όλων όσων ε, συμμετέχουν και εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, θεωρούμε ότι η Επιτροπή στην αξιολόγηση αντικτύπου που έκανε έδειξε με σαφήνεια ότι οι συμβαλόμενοι πρέπει να έχουν κάποια ευελιξία Αλλιώς δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη των καθυστερημένων πληρωμών. Η προθεσμία τα 30, 30 ημέρες, μετά την οποία αυτόματα ξεκινάει η διαδικασία, ιδιαίτερα αν προηγουμένως δεν έχει υπάρξει μια προθεσμία 30 συμπληρωματικών ημερών μετά από διευθέτηση και από διακανονισμό όσον αφορά ε, την πρώτη καταβολή που πρέπει να γίνει το αργότερο. Καταρχά καταρχάς να σεβαστούμε αυτές τις 30 μέρες. Αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό και δεν ε, αναφέρω το όνομα στην οδηγία του 2000, είναι ότι 5-6 χώρες ήδη προβλέπουν αυτές τις 30 μέρες. Εάν αλλάξουν αυτές οι προθεσμίες, τότε και οι εθνικές συνήθειες θα έπρεπε να αλλάξουν. Εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με τις 30 μέρες ίσως, ειδικέ συμφωνίες, εξαιρετικές περιπτώσεις. Αλλά νομίζω ότι οι 30 μέρες είναι μια σωστή προθεσμία, καλή προθεσμία. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, με τα νοσοκομεία. Αυτές τις ταγμούς σας τους κατανοώ, ούτε κι εγώ είμαι ενθουσιασμένη απόλυτα γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είδαμε αυτή την κατάσταση και στην Ανατολική Ευρώπη, στην Νότια Ευρώπη και να υπάρχουν περισσότερα περιθώρια λιγμών στα νοσοκομεία, όχι τόσο για τις προμήθειες για τις οποίες ε, μιλήσατε εσείς, αλλά και για προμήθειες ε, φάρμακων ε, που εξαρτώνται από πληρωμές και κρατικές επίσης προμήθειες. Άρα λοιπόν τα νοσοκομεία εξαρτώνται και από άλλες πηγές. Εύχομαι στις τροπολογίες αυτές να μην ξεχνούμε και αυτούς που σεβάστηκαν τον νόμο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το έκαναν και χάρη σε αυτό άλλωστε συνεχίζουν να είναι παρούσες στην εσωτερική αγορά και στην παγκόσμια αγορά. Γι' αυτό θα πρέπει αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσπαθήσουμε να τις βοηθήσουμε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι ο στόχος όπως την Επιτροπή και για μα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι κάναμε, σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο, ότι έχουμε πολύ λογικές, ε, λογικούς συμβιβασμούς που δρομολογούνται. Προχωρούμε λοιπόν καλά. Να θυμίσω σε όλους την προθεσμία για τις ε, τροπολογίες που είναι η Δευτέρα Μαρτίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Βάιλερ για τη δουλειά σας. Πριν να κλείσω την συνεδρίασή μας, να κάνω κάποιες ανακοινώσεις για τα πρακτικά. Καταρχήν για την ε, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας του κ. Τρατσκόφσκη για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την ε, Ελβετία και τα εμπόδια στην ε, πραγματοποίηση της ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς. Θα ήθελα να παραταθεί η προθεσμία για αυτήν την έκθεση. 8 Απριλίου θα την ξανα